Ξεκινούμε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι στη διάθεσή σας. Σε περίπτωση που δεν εκφραστούν ενστάσεις οι προτάσεις για προσθήκη εγκρίνονται τα Και τώρα θα περάσουμε